Guten Morgen, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σήμερα έχουμε πολύ περισσότερα μέλη παρόντα από ό,τι χθε το απόγευμα. Αλλά τώρα πια φτάσαμε στην Τρίτη το πρωί, δεν είναι Δευτέρα απόγευμα. Καλώς ήρθατε όλοι λοιπόν στη μαραθώνια συνεδρίαση που μας περιμένει με ψηφοφορίες επισημαντικών φακέλων που εξετάσαμε και σήμερα θα αποφασίσουμε εδώ στην Επιτροπή. Ελπίζω ότι όλοι έχετε τις κάρτες σας, τις ηλεκτρονικές για να ψηφίσετε, γιατί πάντα χρειάζεται ένας ηλεκτρονικός έλεγχος. Λοιπόν, να ε, τοποθετήσετε τις ε, κάρτες στην ισοχή ή ε, έχετε τις έτοιμες. Πάμε στο σημείο 10 της σημερινής διάταξης. Η διεθνή εμπορική πολιτική στο πλαίσιο των επιταγών της αλλαγής του κλίματος. Γνωμοδότηση που συνέταξα εγώ, έχουμε 33 τροπολογίες, θα ψηφίσουμε. Τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 2 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τρία Πέρας. 32 προς 17 σαφής οι συσχετισμοί. 4 υπέρ. Κατά αποχές 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Γιολάντα Εμίλια Χίμπνερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ελέγχουμε την 18 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας Απορρίφθηκε. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δέκτη. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 21. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 22 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24. Τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή Περνάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 49 υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές. Το ψήφισμα έγινε δεκτό με μεγάλη πλειοψηφία και θα πάει στην ε, Επιτροπή Εμπορίου που θα ψηφίσει αύριο ο συνάδελφος Περέλο. Θα ήθελα παρακαλέσω, σας παρακαλέσω Πρόεδρε να σημειώσετε στην τροπολογία 3 ψήφισα υπέρ. Δεν δούλεψε το μηχανήμα μου. Ε, είχα βάλει ανάποδα, βλέπετε, την κάρτα μέσα. Είμαι υπέρ της ε, τροπολογίας 3. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χρειάζεστε ακόμα την ε, κάρτα σας. Εντάξει. ευχαριστώ για την υπόδειξη, για την τροπολογία 3. Αυτή ήταν η πρώτη ψηφοφορία και προχωράμε με το επόμενο μέτρο, το 11, για τις έρευνες για πετρέλαιο και την εξόριξη πετρελαίου στην Ευρώπη. Και εδώ υπάρχει ολόκληρη σειρά τροπολογιών. Αρχίζουμε με την 8, Ρίτσαρτ Ζέμπερ Πέτερ Λίζε, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 19. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Προφορική τροπολογία στο πρωτότυπο κείμενο. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Πα. Μαζί. 29-31. Ψηφίστηκαν μαζί. Ναι. Ε, 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 37 Βάις Γκέρμπερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ελέγχουμε την 36. Απορρίφθηκε. Ε, ε, ε, ναι, ναι, ε, δεν το πρόσεξε. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 36 υπέρ. 38 κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 και 41 από κοινού υπέρ όχι όχι χωριστά τη 40 πρώτα τη 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 υπέρ. Κατά. Ποχές δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Αυτά ήταν οι τροπολογίες. Ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία άρχεται. 46 υπέρ 8 κατά 3 αποχές συγχαρητήρια στους συντάκτες της γνωμοδότησης για την ε, εξόρυξη πετρελαίου στην Ευρώπη. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και πάμε στο σημείο 12. Σημείο 12. Έκθεση Μάρτιν Κάλαναν. Πρότυπα εκπομπών για τις επιδόσεις των καινούριων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Ist die Prozedur? Διαδικαστική πρόταση από τη Ρεμπέκα Χάρμς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι η ομάδα μου ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για τις εξής ε, ενοποιημένη τροπολογία 1 που ψηφίζεται μαζί με, την ενο... με το ενοποιημένες 2 και 3, την ενοποιημένη 9 που ψηφίζεται μαζί με την ενοποιημένη 10, την ενοποιημένη 5 που ψηφίστηκε, ψηφίζεται με την 6 ενοποιημένη, την ενοποιημένη 4 και όλες τις τροπολογίες στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, έχει κατατεθεί η πρόταση των Πρασίνων για ονομαστική ψηφοφορία ε, σύμφωνα με την διαδικασία, αν συμφωνούν όλοι και τους, ε, τον κανονισμό, αν συμφωνούν όλοι εντάξει, αν το 1 τέταρτο των ε, βουλευτών διαφωνεί, τότε δεν γίνεται. Όχι, το αντίθετο ισχύει. Υπάρχει δικαίωμα της μειοψηφία. Αν ένα τέταρτο των μελών ενίστανται, 16 δηλαδή εν προκειμένου, τότε το σημείο αυτό θα ψηφιστεί ηλεκτρονικά. Θα ψηφιστεί ποιος είναι υπέρ της ονομαστική ονομαστικής ψηφοφορίας με... πάνω στα θέματα αυτά που ακούσατε. Okay, sind also weit mehr als 16. Äh, Είναι πολύ περισσότεροι από 16. Ο καθένας το βλέπει. Λοιπόν, Ρεμπέκα, δεν το έχω στον κατάλογο, θα προσέχομαι, αλλά να έχεις, να έχεις στο νου σου, μήπως και ξεχάσουμε να ψηφίσουμε καμία ηλεκτρονικά. Αρχίζουμε. Είναι μακρά η ψηφοφορία. Μέχρι ήρθε και ο Έλμαρ Μπρόκ για τα ελαφρά επαγγελματικά, ε. Ενδιαφέρον αυτό. Καλώς τον. Λοιπόν, αρχίζομαι. Ήτρε 1. Κρίς Ντέιβις. Ο κύριος Μπρόκ ήξερε ότι αυτή είναι Επιτροπή Περιβάλλοντος. Στα 10 χρόνια τον έχω ματαδεί. Ευπρόσδεκτος όμως likes to vote... Uh, ναι, ο βαρέων βαρών θέλει να ψηφίζει για ελαφρά ζητήματα. Ε, θέμα πολιτική ανθρώπων κλπ. Συγγνώμη για τα σχόλια. Λοιπόν, συγγνώμη για το σχόλιο. Αρχίζουμε. Τροπολογία Ήτρε 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στις ενοποιημένες ε, τροπολογία 1, εδώ θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται. warten, bis der Kollege να περιμένουμε με τις κάρτες πέρα της ψηφοφορίας. 23 υπέρ 36 κατά μία αποχή απορρίφθηκε. Άρθρο 1. Παράγραφος 1. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56, 57, 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 60 υπέρ. κατά αποχές δεκτή. Τώρα, ενοποιημένη τροπολογία 9, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 32 υπέρ 27 κατά μία αποχή δεκτή. Λοιπόν, η τεχνολογία λειτουργεί, εντάξει είναι το αποτέλεσμα. Πάμε στη σελίδα 3. Στην 74. Βάις Γκέρμπερ Γκροστέτ κλπ. Υπέρ. 74. Αυτή ψηφίζουμε. Κατά. Αποχές. έλεγχος ηλεκτρονικός ζητήθηκε άλλωστε. Πέρας. «29 υπέρ 31 κατά». Απορρίφθηκε λοιπόν. «75 υπέρ». ονομαστική πάλι. Όχι. Υπέρ, υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίφθηκε. Ήτρε 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 78, 79, 80, 81. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76-77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Ήτρε 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δέκτη. Τραν υπέρ κατά αποχές δεκτή 383 τραν 8 ήτρε 14 υπέρ κατά αποχές δεκτές 84 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ελέγχουμε την 84. Πλευράς. Απορρίφθηκε. Ήτρε 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 85. 88, 91, 93, τραν 10, ήτρα 16, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 86-92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 89 ήτρε 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή, δεκτές. 87, 90, 94, τραν 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Όχι. Είμαστε στην 87, 90, 94 και τραν 9. Επανάληψη ψηφοφορίας. Υπέρ παρακαλώ αυτών των τεσσάρων. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Έτσι. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 και 104. 99 και 104 υπέρ. Α, είναι δύο διαφορετικές. Είναι περίεργο. Μόνο, μόνο την 99 ψηφίζουμε. Δεν είναι καλά παρουσιασμένα. Υπέρ της 99. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104 τώρα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98, 100, 101, 102 και 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτονται. 97 ήτρε 18 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορριπτονται. Έλεγχος. Πέρασης ψηφοφορίας. Απορρίπτονται έτσι δεν είναι. 95. Γκρότε υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η τραν 11 καταπίπτει. Και πάμε στην ενοποιημένη τροπολογία 4 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. <clears throat> Πέρας. 25 υπέρ 37 κατά. Απορρίφθηκε. 105 βίλς υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 18 Μπερλάτο 111 108 υπέρ όλα μαζί κατά αποχές απορρίπτονται η κυρία Πέρσκα θέλει έλεγχο έλεγχουμε λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίφθηκαν. Η, η πλειοψηφία. Τώρα, 109-110 σε υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. 115 ή 318 ίδιες ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. 114 υπέρ. Α, και 117 πάνε μαζί υπέρ. 114-117 ψηφίζουμε για τις δύο. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτονται. 112 και 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τραν 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113 Αντωνέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Α, θέλει έλεγχο κυρία Βάις Γκέρμπερ. Ψηφίζουμε την 113. Άρχεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Ε, περισσεύει μία ψήφος του ΕΛΚ, πρέπει μια κάρτα να αφαιρεθεί. Βγάλτε μία κάρτα από το ΕΛΚΑ. Εξακολουθεί να περισσεύει μία. Πέρας. Τώρα ήταν εντάξει. Απορρίφθηκε. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 119-120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 124-127 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Α, ήταν μέσα σε αυτή την κατηγορία και το ΙΤΡΑ 18. Και συνεχίζουμε με 123 και 126 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτονται 121 και 128 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται 122 και τραν 12 υπέρ. 122 τραν 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 130-131 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 132, 133, 134 Γκαρντίνι Βαλεάν Μπερλάτο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται 136 ήτρε 18 141 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 138 και 140 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές έλεγχος και ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες έχουν μια περισσευούμενη εξακολουθούν να έχουν μία παραπάνω. Τώρα είναι εντάξει. Πέρασε της πληροφορίας. Δέκτη. νοποιημένη τροπολογία 15. Ψηφίζεται όσο έχει υπέρ. Κατά. Αποχές. Τι θα έλεγα εγώ. Έλεγχος. Έλεγχος. Θα το δούμε. Περισσεύει μια ψήφος σοσιαλιστών δημοκρατών. Πέρας. Ναι, ήταν σαφές 37 προς 25 δεκτή. Τώρα θα πάμε στη σελίδα 11, 142, 100... μέχρι την 143. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ενοποιημένη 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Νομίζω ότι ήταν σαφές, αλλά θα ελέγξουμε την 13. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία, ενοποιημένη 13. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίφθηκε λοιπόν. Τυχερός ήμουνα. Φάνηκε ότι ήταν σαφές, αλλά καμιά φορά δεν είναι τόσο. Εκατόν σαράντα τέσσερα, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ταυτόσημη με 150-151 απορρίφθηκαν. Τραν 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 152-153-154. υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Άρχεται η ψηφοφορία, ελέγχουμε για αυτές. Πέρασε. Απορρίφθηκαν. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία 14. Ψηφίζουμε κανονικά υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρ. Α, τη 14 να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δύσκολα να δεχτεί κανείς τις ήτες, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτές. Απορρίφθηκε. Η 158 στο άρθρο 5, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 19, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 160 υπέρ. Ήτρε 19 έγινε δεκτή. Α, όχι, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ήτρε 19. Πέρας. Δεκτή. Και τώρα καταπίπτουν μερικές. Ε, πάμε ούτσι και 162 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 163-159 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Απορρίφθηκαν. Ήτρε 19 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 165 Όχι, πάμε στο Inden 3, γιατί έχουμε δεχτεί τιμή. Inden 3, 166-167, παύλα 3 δηλαδή, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 169 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 163 και 159 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Ήταν μέσα και η τραν 18, οπότε συνεχίζουμε με την 163-159. Μισό λεπτό. Την τραν 18 δεύτερο τμήμα θα την ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 163 και 159 είναι ταυτόσιμες και οι 168, Βάις Γκέρμπερ και άλλοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Ήτρα 19, τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεν φαίνεται. Θα ελέγξουμε. Ήτρα 19. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Δεκτή. Συνεχίζουμε. Ήτρα 19. Τέταρτο τμήμα και Αντωνέσκου 171 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ μαζί με τις άλλες. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Ενοποιημένη τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. έλεγχος. Ενοποιημένη 7. Πέρας. Για να ξέρουν όλοι τις, τους συσχετισμούς. Απορριφθήκε. 146 και 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Ήτρε 20-148 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές δεκτή ενοποιημένη τροπολογία 16 και η 7 του εισηγητή μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Ενοποιημένη τροπολογία 17 συν την 8 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Ενοποιημένη τροπολογία 18 μαζί με την 9 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή άρθρο 7 τροπολογία 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 173, 176 και ήτρα 21 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 174 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 179 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, την 177 εννοούσε. 178, 179 ή 32 μαζί. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά. ...182. Υπέρ πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 183, 181 Ήτρα 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 187, 188 Ήτρα 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 8 κανονική ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές δεκτή 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 190, 91, 192 ή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτές 172 υπέρ κατά αποχές δεκτή 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 193 πρώτο τμήμα, 194 πρώτο τμήμα, 195 ή 326 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τραν 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193 δεύτερο τμήμα, 194 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 198 πρώτο τμήμα, 199 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται, άρθρο 8, 200 και 203 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά ε, αποχές απορρίπτεται ήτρα 21 υπέρ 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ενοποιημένη τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Επόμενη σελίδα. 211, 212, 199, 213, 198, δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 214, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 215, 216, 217 198, 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 219, 220, 221, 222 και 198 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ενοποιημένη τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή επόμενη σελίδα ενοποιημένη τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τραν 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 229 πρώτο τμήμα και 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 μαζί με 229 και 231 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 232-233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τραν 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 236-237 Ήτρε 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 239 Ήτρε 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 238-240 υπέρ κατά αποχές δεκτές 234 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Η 234. Η πράσινη έχουν μια περισεβούμενη κάρτα ποτέ δεν είναι αρκετέ, ποτέ δεν είναι υπερβολικά πολλέ. Λοιπόν, τέλο πέρα Ε, δεκτή. 33 προς 29. Δεκτή. Τραν 25 ή 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τραν 26 ή 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Ήτρε 31 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Του εισηγητή 13 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει γιατί έγινε δεκτή το 31 ήτρε. Πάμε στη συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ενοποιημένη τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Απορρίπτεται. Α, ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλεγχος. Πέρας. Εκπληκτικό. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη 241 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 242 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος στη 242. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πραγματικά παραμισή τρίχα, αλλά απερίφθη. 243, 244, 245, τράν 28, ήτρα 32. Υπέρ. κατά. Αποχές δεκτές. Ενοποιημένη τροπολογία 22. Μαζί με τη 246 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 247 υπέρ. Ζητείτε έλεγχο στην 22 ενοποιημένη και τη 246. Πέρας λοιπόν. Απερίφθη όντως, απερίφθησαν. Εντάξει, 247, λεπάζ, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 248 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τραν 29 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 33 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία 10 Η 10 ήδη έχει γίνει δεκτή μέσω προηγούμενης ψηφοφορίας που εκάμαμε ε, όταν ψηφίζαμε την ενοποιημένη 9. Σύμφωνη. όλοι. Πάμε στην ενοποιημένη 6 λοιπόν. Αυτή καταπίπτει όμως. Και έτσι Πάμε στη σελίδα 27, γιατί όλα τα άλλα καταπίπτουν. Σλίτερ Χάρμς 266. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 228, 268 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 270-269 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 271 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 273 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 274, 275, 276 υπέρ. Καταπίπτει, α, Καταπίπτουν. Μάλιστα. Η 33, καταπίπτει και αυτή. Συμβιβαστική 11, υπέρ. Της 11 συμβιβαστικής τροπολογίας. Κατά. Αποχές

κατά αποχές απορρίπτεται 282, 283 και 251 και 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβιβαστική 12 και 284 υπέρ κατά αποχές δεκτές. Ενοποιημένη τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 12 παράγραφος Τέλο πάντων, η τροπολογία 285 μαζί με τη 286, 288 και 289. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Δεκαπέντε. Λοιπόν, στη 15 θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Πάλι, ποιο είναι κατά. Αποχές. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Αν θέλετε μπορούμε να ελέγξουμε. Το 15 πρώτο τμήμα, αν θέλετε, έλεγχος ηλεκτρονικός. Δεκτό. 287 ήτρε 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Όχι, όχι, όχι. Οι δυο αυτές καταπίπτουν. Ναι, ε, προχωρούμε με τη συμβιβαστική 7 κατά αποχές δεκτή η 290 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Η 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στα παραρτήματα. Ήτρε 35 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. Δεκτή. 291 υπέρ. Όχι, όχι, καταπίπτει. Καταπίπτει. Τώρα θα συνεχίσουμε στην ενοποιημένη 2, με την ενοποιημένη τροπολογία 2. Έτσι δεν είναι. Υπέρ. Τροπο... Ε, ενοποιημένη 2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 295 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 294 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 296 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ενοποιημένη τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήτρε 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 298. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 35. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 299 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 301-302 υπέρ κατά αποχές δεκτές 303 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Έλεγχος της, της 303. Πέρας. Έχει απορριφθεί λοιπόν η 303. 304. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 305-306 υπέρ. Α, και η ΙΤΡ 37 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 307 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 308-309 τραν 32 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 310 υπέρα Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος την 310. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μετά πάμε στις, στα recital, τη 17 υπέρ. κατά τις 17. Όχι, μισό λεπτό. Ε, ε, ψηφίζουμε 17 πάλι. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 2, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 και ήτρε 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται απορρίπτονται. Ενοποιημένη τροπολογία 20 και 21 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ήτρε 4 υπέρ. κατά αποχές έλεγχος, ελέγχουμε την Ήτρα 4. Πέρασε Δεκτή. Πάμε στην 24 και στην 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Η 26 καταπίπτει και 27 καταπίπτει. 28. Ποιος είναι υπέρ της 28. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 30, 31, 33 και ίτρε 5 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτονται. 32 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36, 37, 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τραν 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 41, 44 και ήτρα 7 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, 46 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 45 υπέρ. Ποιητικά είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Τραν 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τραν 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή ήτρε 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή ήτρε 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 και 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 10 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, ελέγχουμε. Την Ήτρε 10. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τραν 5 και 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορριφθήσαν 52 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές δεκτή και συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ματίας, ζητώ να κάνουμε μία διακοπή πριν πέντε λεπτά διακοπή πριν πάμε στην τελική ψηφοφορία. Μάλιστα, γιατί και εμείς θέλαμε να ελέγξουμε, μπας και ξεχάσαμε τίποτα. Ε, πεντάλεπτο διάλειμμα. Seid ihr Είστε όλοι εδώ, ναι. Ähm, λοιπόν, πριν προχωρήσουμε και πάμε στη τελική ψηφοφορία, έχουμε τρεις τροπολογίες που μας ξέφυγαν. Λοιπόν, σας παρακαλώ, πηγαίνετε στη σελίδα 30. Στα παραρτήματα τα οποία είπαμε ότι τα είχαμε τελειώσει αλλά δεν τα τελειώσαμε γιατί δεν έγινε δεκτή η, ενοποιημένη τέσσερα σελίδα 30, 291, 292 και ήτρε 35, δεύτερο τμήμα. Αυτές τις τρεις πρέπει να ψηφίσουμε πριν περάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Στη σελίδα 30. 291 Βίλς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 292 υπέρ Σβάις Γκέρμπερ κατά αποχές απορρίπτεται και ήτρε έλεγχος Έλεγχος στις 292 λοιπόν. Πέρας της ψηφοφορίας, όντως απερίφθη, και ήτρε 35 δεύτερο τμήμα υπέρ Κατά. Αποχές απερίφθη επίσης. Οπότε εντάξει. Τώρα είμαστε εντάξει. Τα ψηφίσαμε όλα όπως έπρεπε και πάμε στην ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία. Ναι. Ονομαστική ψηφοφορία. 31 υπέρ, 25 κατά, 2 αποχές. Και η δεύτερη ψηφοφορία για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 32 υπέρ 25 κατά μία αποχή ε, συγχαρητήρια στον εισηγητή Μάρτιν Κάλαναν. Ο εισηγητής ζητεί το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, δεν ήμουν εδώ στην ψηφορία για το σχέδιο της ε, έκδοσης. Εγκρίθηκε. Δεν την είδα στην οθόνη. Μπορείτε να μου πείτε τα αποτελέσματα. Πριν φύγει ο κόσμος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χιώδεις εισηγητές. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη επίπονη διαδικασία. Δεν τα βρήκαμε με συμβαστικές ε, τροπολογίες, γι' αυτό και είχαμε αυτές τις, ε, ενοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά τους ευχαριστώ όλους. Ε, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, ελπίζω να συνεχιστεί καλή συνεργασία Είχαμε πολιτικές διαφορές σε επίπεδο πολιτικών ε, απόψεων, αλλά ε, επί του προσωπικού τα πήγαμε τέλεια. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ και εγώ του Κιώδης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 31-25-2. Το πρώτο. Και το άλλο ήταν, ναι, 58, πάει 32-25-1. Το τελευταίο για το νομοθετικό ψήφισμα. Επόμενο, το 13. πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή τροποποίηση του κανονισμού 726 του 2004. Κρίστοφερ Φιέλνερ. No, Είχε ανοίξει το μικρόφωνο ο μιλητής. Oh, Α, είχα ανοίξει, αλλά ήταν το λάθος μικρόφωνο. Ξέρω ότι πιέζει πάρα πολύ ο χρόνο. Οπότε γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό το πόσο υπήρξε πρόθεση του, να συμβαστούμε, γιατί αν πριν από ένα χρόνο ε, έλεγε κανεί σε ποια φάση θα βρεθούμε σήμερα, τότε θα ήταν απίστευτο. Κανεί δεν θα πίστευε ότι θα υπήρχε τόσο ευρεία συνένεση για όλα αυτά όπω και έγινε και, για τι συμβαστικέ και για τι ενοποιημένε τροπολογίε. Και τελικά το καταφέρω τόσο εγώ όσο το πόσο επικοδομητικοί ήσαντε οι σκιώδεις συγκητές. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Dank für... Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ όλους που συνεργάστηκαν. Σιλβανιό. Oui, Monsieur le Président, quelques mots. Euh. Δύο λόγια ταχαίως κύριε Πρόεδρε. Ε, σε συνέχεια των όσων μας είπε ο κύριος Γέλνερ, ο εισηγητής μας, όντως ε, έτσι προχωρήσαμε ε, ικανοποιητικά για την σύνταξη αυτών των δύο κειμένων και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έτσι τα καταφέραμε. Βεβαίω υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία προστριβής και θα δούμε τι θα γίνει στις ψηφοφορίες. Έχουμε και τα συμβεστικά ένα και δύο Ακόμα ε, δεν τα έχουμε βρει, αλλά πέραν αυτών τα καταφέραμε να απαλύνουμε τις διαφορές μας και έτσι να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση. Ε, Ο Κάρλ Σλούτερ για την τροπολογία. Ναι, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή, παλιοικοδομητικά. Τα πήγαμε σε αυτή τη διαδικασία, υπήρξε διάλογο και γι' αυτό και εγώ τώρα αποσύρω την τροπολογία μου, την υπαριθμόν 3, διότι η αρχική πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρήσαμε ότι δεν θα αποδώσει όμω λόγω τη καλή πίστη του εισηγητή. Τώρα καταλήξαμε σε κάποια πρόταση που μπορεί να είναι αφετηρία να δουλέψουμε και επομένω για την απόρριψη, την τροπολογία, τη σχετική, την αποσύρω. Το νούμερο 3. Uh, Αρχίζουμε λοιπόν. Τροπολογίες 6 και 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκαν. 8 και 9. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίφθηκαν. 10 και 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 13 υπέρ. Τα, ταυτόσημη. Υπέρ. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 13-14 ήταν μαζί. Πάμε στην ΙΜΚΟ 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. ΙΜΚΟ 4. Υπέρ. Κατά. ΙΜΚΟ. ΙΜΚΟ. Όχι ΙΤΡΕ 4. ΙΜΚΟ 4. Η άλλη κατέπεσε, γιατί ήτρε. Ήμκο 4, υπέρ, ξανά. Ήμκο 4. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος. Έλεγχος στις 2. Πέρας. Οι δύο λοιπόν απορρίπτεται. 15-16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτές. Ήμκο 5 και Ήτρε, η Ήτρε 5 ε, καταπίπτει. Η 15 υπέρ. Α, η πρώτη καταπίπτει 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ήμκο 7 ή τρεπτά, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε 20-21 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 22 υπέρ. κατά αποχές απερίφθη ήτρε 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 8 καταπίπτει 23 σλούτερ υπέρ κατά αποχές απερίφθη 24 υπέρ Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Α, ελέγχουμε την 24 κατόπιν επιθυμίας του. Εντάξει. Πέρασε. Απερίφθη. Οι φιλελεύθεροι ψηφίζουν μέσω του συντονιστού τους. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη επίσης. Τώρα, στα recital. Ήμκο 1, ήτρα 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Ένα του εισηγητή υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΤΡΕ 2 κατά πίπτη αυτή μετά 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε ΙΤΡΕ 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 52 υπέρ 2 κατά 3 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για το εγχείρημα αυτό. Ακούω ότι πρέπει να κάνουμε και δεύτερη ε, τελική ψηφοφορία γιατί είναι νομοθετικού περιεχομένου. Οπότε ψηφίζομαι το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 51 υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές. Και πάλι συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα πάμε στο 14, την οδηγία δηλαδή, Αυτή τώρα είναι μεγάλη ψηφοφορία όπως βλέπετε κι εσείς. Τον ίδιο λόγο όπως και την προηγούμενη έκθεση και εδώ αποσύρουμε την τροπολογία μας για απόρριψη για τους ίδιους λόγους. Λοιπόν, πάμε στη σελίδα 2 και στο άρθρο 1. Συμβιβαστική ένα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική δύο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ενοποιημένη τροπολογία ένα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ενοποιημένη δύο υπέρ. Κατά. Αποχές Έλεγχος. Πέρας. Απερίφθη. Ενοποιημένη τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ενοποιημένη τροπολογία 4. Υπέρ κατά αποχές δεκτή ενοποιημένη τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 82. Πρώτο τμήμα ψηφίζεται υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Ήμκο 11. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 83 με τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ήμκο 12 ήτρα 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθησαν. 84 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθησαν. 86 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 87 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 88, 89 και ήτρο 8 υπέρ κατά αποχές δεκτές 90 υπέρ κατά αποχές δεκτή 91 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 97 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 96 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. «98. Ζήλ Παρνιό. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 99 και 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 102 υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Επόμενη σελίδα. 110. Κάρλ Σλούτερ υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 12. Α, έλεγχος. Ναι, την 110 να ελέγξουμε. Πέρας. Δεκτή. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Επόμενη σελίδα. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήμκο 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 119 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 16. Α, έλεγχος της 119. Μάλιστα. Δεν εμπιστεύεστε τον Κάρλ Σλίτερ. Πέρασε. Δεκτή. Ήμκο 16 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Όλες οι υπόλοιπες πρέπει να ψηφιστούν. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Έλεγχος της 120. Πέρας. Δεκτή. 121-122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 121-122 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Δεκτές. Ήτρε 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 123-124 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 125 υπέρ. Α, καταπίπτει αυτή. Ναι, σωστά. Επόμενη σελίδα. 126 και ίνκο 18. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 127 και ΙΜΚΟ 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθησαν. 13. Α, έλεγχος 127 και ΙΜΚΟ 19. 13 Δεκατρία εισηγητή. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ο κατάλογος των ψηφοφοριών λέει ότι η τροπολογία 129 καταπίπτει αν εγκριθεί η ενοποιημένη τρία και καλύπτεται από αυτήν. Όμως εδώ το θέμα είναι ποιες πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται και η τροπολογία 9 πάει λίγο πιο πέρα και προσθέτει κάτι εδώ και μπορεί να γίνει δεκτή ως προσθήκη μετά το άρθρο 1.5 σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν και θέλω να το διαβάσω ε, προστίθεται και ένα ε, κοιτίο πληροφοριών με πληροφορίες, με ευανάγνωστα ορατά στοιχεία διαφοροποιημένα από το υπόλοιπο κείμενο. Αυτό το κουτάκι περιλαμβάνει το πεδίο, περιγράφει σύντομα τις ενδείξεις για το φάρμακο, ούτως ώστε να κατανοήσει ο ασθενής τα υπέρ και τους και να το παίρνει με ασφάλεια το φάρμακο. Νομίζω ότι μπορούμε την προσθήκη αυτή να την εγκρίνουμε και ρωτώ τον εισηγητή εάν συμφωνεί. Εδώ το Προεδρείο λέει ότι καλύπτεται το θέμα αυτό από την ενοποιημένη τρία και θα δημιουργήσουμε πρόβλημα αν ξαναψηφίσουμε. Μάλλον ε, τίνω να πω ότι δεν θα το ψηφίσουμε γιατί έχει ήδη καλυφθεί. Καλύπτεται. 128. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Καταπίπτουν όλα αυτά. Όλες καταπίπτουν αυτές. Αυτό είναι το μαγικό που μας έκανε η προηγούμενη ψηφοφορία. Θαυμασία. Λοιπόν, σελίδα 15 πάμε. 187 Ζιλ Παρνιό. Υπέρ. Ζιλ. Αποσύρθηκε η τροπολογία, πρόεδρε. So, Και αυτή λοιπόν και η 187 έχει αυτό και η 188 έχει αποσυρθεί, οπότε πάμε στην ΙΜΚΟ 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. ή 23. Ήτρα 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 189 ήμκο 32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Ήτρα 24 γλωσσική και Ήτρα 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Ήτρα 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρα 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 196 και ΙΜΚΟ 33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. «197 Μαρίνα Γιανακουδάκη. Υπέρ». «Κατά» αποχές δεκτή. Ήτρα 29 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 198-199-200 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Ήτρα 30 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήτρο 30 ελέγχουμε. Γιατί. Ψήφισαν όλοι. Υπέρ, ναι. Ο εισηγητή πάντω ήταν υπέρ, ναι, σωστό είναι αυτό. 201 ε, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 205, 206, 207 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Ήμικο 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18-209 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 210 και ΙΜΚΟ 35 υπέρ κατά αποχές δεκτές 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 212 υπέρ κατά αποχές δεκτή 217 υπέρ κατά αποχές Διακόσια 223-224 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 225-226 υπέρ, κατά αποχές δεκτές 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ...228 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, ήτρε 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 229-230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 20 ή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή ήτρε 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή Πέτα Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ την 231 να την ψηφίσουμε τμήματικά. Στο δεύτερο τμήμα να αρχίσουμε εκεί που λέει by way of derogation μέχρι το τέλος του κειμένου. Να ψηφίσουμε χωριστά το πρώτο τμήμα. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση θα το θέλαμε πολύ και ευχαριστούμε. Υπάρχει ένσταση κατά της τμηματικής ψηφοφορίας. Όχι. Εντάξει. Ψηφίζουμε λοιπόν, εφόσον όλοι γνωρίζετε τι ψηφίζετε. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό το πρώτο τμήμα. Πάμε στο δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Και αυτό δεκτό. 2.33. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 236-237 υπέρ κατά αποχές Λέω ναι, εγκρίνεται, αλλά θα το ελέγξουμε. Πέρας. Όχι, άξιζε τον κόπο που το τσεκάραμε γιατί απερίφθησαν. Ε, φαίνονται αυτά, κυρία Σνέλχαρτ. 2.38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.39, 2.40, 2.41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 2.42 υπέρ. Όχι, 244. Ε, απερίφθη. Το 244 απερίφθη, 245. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.47 ήμικο 38 υπέρ κατά αποχές δεκτές 2.48 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ήτερ 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 39 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 τμήματικά. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Πάμε στην επόμενη σελίδα. Είμαι 42 και 267 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 268 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 273 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 2,72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 271 και ΙΜΚΟ 43 υπέρ. In... Α, υπάρχει ένας υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή, είπε. Ή 38, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 274, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2,75 υπέρ. αποχες αποχές δεκτή 277-278 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε τις 277-278. Εγκρίθηκαν. Και πάμε τώρα στη 280, Κορίν Λεπάζ, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 283, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην επόμενη σελίδα. 285. Γύριμα στάλκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 286. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήτρε 40 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 287 και ΙΜΚΟ 45 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 291 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ήτρε Δεκτή. 42 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 2,94. Α, είναι ταυτόσιμες. Καλά. 24. Με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 25 υπέρ. Ε, κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ κατά εποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 295 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή και πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις recital 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 και ήμκο 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30. Τμηματική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό και δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές δεκτό 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή ήτρε 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 και ΙΜΚΟ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 44-45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Επόμενη σελίδα. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 56 Πρώτο τμήμα υπέρ. Νέσα Childers υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στην 5 μόνο το πρώτο τμήμα πάλι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 55 ούτσκι υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, ήτρε τρία καταπίπτη εξήντα ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ήμκο 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και πάμε στην τελευταία σελίδα τι τύχη ήταν αυτή. Ήτρε 6. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ήτρε 6. Πέρας. Απερίφθη. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ίνκο 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή Και πάμε στην τελική ψηφοφορία. Επί του σχεδίου εκθέσεως όσο τροποποιήθη. Άρχεται η ψηφοφορία. να πατήσει το κουμπάκι του και ο συνάδελφος Σόνικ. Ψηφίσατε. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. 48 υπέρ, μία ψήφος κατά, τρεις αποχές και δεύτερη ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Νομοθετική, ε, άρχεται ψηφοφορία.